Okay. This year, there's been one year since the... Πέρασε ένα χρόνος από το κίνημα MeToo. Θα σας πω μερικά γεγονότα. Μετά το κίνημα αυτό, γιατί εγώ ασχολήθηκα από την αρχή, έγιναν μια-δυο προτάσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ξαναπάνε οι πολιτικοί στο σχολείο, να κάτσουν στα πρανία και να τους διδάξουμε το θέμα της παρενόχλησης. Υπήρχε ένα σχέδιο για εκπαιδευτικά σεμινάρια και διασκέψεις όπου οι πολιτικοί που ασχολούνται με καθημερινά θέματα, με παιχνίδια γύρω από τους μισθούς ανδρών και γυναικών, ε, ε σχόλια ύπουλα, ύποπτα, συκοφαντικά ας πούμε στο, στα γραφεία και από τους 751 ευρωβουλευτές μόνο 32 βουλευτές ήθελαν να ε, κάνουν αυτά τα σεμινάρια. Ε, θέλω να ρωτήσω τους υπόλοιπους γιατί δεν θέλουν να πάνε σε αυτά τα μαθήματα. Και τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνιών ε, και εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα σας πω, θα μας κάνει κάποια εισαγωγικά. Ευχαριστώ, Τερέζα. Σας ευχαριστώ όλους που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθετε σε αυτό το σεμινάριο σήμερα τύπου που οργανώνεται στα πλαίσια της Διεθνούς ημέρας για τη γυναίκα. Όταν συζητήσαμε μεταξύ μας και με τα μέλη της ε, Επιτροπής για τα Δικαιώματα Γυναικών, είπαμε ότι είναι ένα σεμινάριο που γίνεται 79 ακριβώς μέρες πριν από τις ευρωεκλογέ. Και επομένως θα πρέπει να εστιάσουμε σε ένα βασικό θέμα που είναι η θέση των γυναικών στην πολιτική και πόσο μπορούμε να υποφεληθούμε από τις επόμενες ευρωεκλογές... ούτως ώστε να ενισχύσουμε το ρόλο, την σημασία των γυναικών στο, στην ευρωπαϊκή πολιτική και πώς μπορούν να συμμετέχουν πιο πολύ σε νούμερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Σήμερα και αύριο θα, ε, θα ενημερωθείτε για όλα όσα έχουν γίνει, όλα τα project, τα εργαλεία, τις πλατφόρμες που έχουμε δημιουργήσει και που διαδίδουμε, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει τη σημασία των επόμενων ευρωεκλογών. Τι παίζεται, τι διακυβεύεται και ποιος θα είναι ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου τα επόμενα πέντε χρόνια. Και γιατί το να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα περισσότερο παρά Είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουμε. Και θα δείτε επίσης αυτό το διήμερο και κάποια άλλα στοιχεία. Ότι η διάσταση του φύλου είναι πολύ πιο έντονη σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Αν συγκρίνουμε με προηγούμενες ε, ευρωεκλογές. Θα δείτε στα προϊόντα μας, στις εικόνες μας, στα μηνύματα που στέλνουμε, ότι κάναμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να περιληφθεί πλήρως η διάσταση του φίλου και η άποψη της γυναίκας ε, στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, στη φρασιολογία που χρησιμοποιούμε και στις στρατηγικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε απέναντι σε τρίτους. Μερικές φορές αυτή η τρίτη φορείς δεν εννοώ ότι είναι πολιτική φορείς, αλλά μιλάω για οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Και αυτοί οι συνομιλητέ ενδιαφέρονται πάρα πολύ να σπρώξουν την, το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Ένα από τα βασικά στοιχεία της προσπάθειας για τις επόμενες εκλογές θα είναι ότι οι δραστηριότητε που οργανώνουμε προσπαθούμε να, τις, να εμπλέξουμε εκεί και άλλους φορείς, οργανώσεις, αλλά και πρόσωπα. Στην περίπτωση των οργανώσεων ε, υπογράφουμε και μάλιστα την τελευταία εβδομάδα υπογράψαμε δεκάδες εταιρικέ σχέσεις με διάφορους φορείς, με διάφορες οργανώσεις και προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε εκείνες τις οργανώσεις που δεν δουλεύουν ε, συγκεκριμένα για τα θέματα των γυναικών, αλλά στα θέματα συναφή ε, με τις γυναίκες και την πολιτική και ειδικά με τις οργανώσεις που ασχολούνται με την ευρωπαϊκή πολιτική. Θα ήθελα να τονίσω το εξή. Ότι το λόμπι για τα δικαιώματα των γυναικών που ζητάει 50% ε, εκπροσώπηση των γυναικών στις ευρωεκλογέ και που θέλει ισότητα απόλυτη στο Ευρωκοινοβούλιο, ισότητα και στους, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 50% γυναίκες, 50% άνδρες επίτροποι δηλαδή, αλλά προσπαθεί να προωθήσει και άλλες ε, θέσεις για τις γυναίκες. Επίσης, μια άλλη οργάνωση ε, που λέγεται Women Political Leaders, γυναίκες ως πολιτικοί ηγέτες ε, ε, και είναι γυναίκες οι, οποίοι έχουν, οι οποίες έχουν φοβερές πολιτικές ευθύνες, είτε για είναι βουλευτές, είτε υπουργοί, είτε αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, συνεργάζονται και κάνουν εκστρατεία ούτως ώστε να προωθήσουν τα γυναικεία θέματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσα να σχολιάσω πολλά άλλα πράγματα μαζί σας για το πώς οργανώνουμε αυτή την εκστρατεία, για το πώς προωθούμε όλα αυτά τα στοιχεία, όλες αυτές τις δράσεις που συνδέονται με το ρόλο των γυναικών στην πολιτική ενόψη των ευρωεκλογών. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ και αν έχουμε χρόνο είτε σήμερα είτε αύριο θα ήθελα οι συνάδελφοί μου να σας μιλήσουν για το τι σημαίνουν οι συνολικές κατευθυντήριες αρχές για την επικοινωνία. Ε, κυκλοφορούν ε, σε όλες τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όταν μιλάμε για την πολιτική του Κοινοβουλίου, για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου, όταν μιλάμε για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα μέλη του Κοινοβουλίου, πάντα έχουμε και μία διάσταση ισχυρή για το θέμα του φίλου. Συνολικές κατευθυντήριες γραμμές για την επικοινωνία λέγονται αυτές. Υπάρχουν πολλά στοιχεία για το πώς θα εφαρμόσουμε την ουδέτερη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα φύλου ε, που υιοθετήθηκε από την ύπατη επιτροπή που προεδρεύεται από τον αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Παπαδημούλη, ούτω ώστε η Ομιλητέ σε διάφορες εκδηλώσεις να έχουν ουδέτερη γλώσσα σε θέματα φύλου. Να αποφύγουμε να έχουμε πανελίστε μόνο άντρες. Ε, επίσης, στην επιλογή των θεμάτων. Ε, στη δουλειά που κάνουμε με τον τύπο. Πώς θα εξασφαλίσουμε ισορροπία στη, στο, στα δύο φύλλα όταν προτείνουμε, ας πούμε, ομιλητές ή καλούμε ομιλητές ή παίρνουμε συνεντεύξεις κτλ. Θέλουμε να υπάρχει μια ισορροπία ε, ως προς το φύλλο. Υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Ε, θα ήθελα να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το έγγραφο όταν σας μοιραστεί, γιατί είμαστε πραγματικά περήφανοι για το γεγονός ότι το υιοθετήσαμε αυτό το έγγραφο και ότι τώρα θα αρχίσουμε να το εφαρμόσουμε πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Σας εύχομαι καλές εργασίες αυτό το διήμερο Πιστεύω θα είναι ενδιαφέρουσα εμπειρία και για από προσωπική άποψη και για τους δημοσιογράφους και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος όχι μόνο είναι ευρωβουλευτής, είναι και αντιπρόεδρος όμως του Κοινοβουλίου και πρόεδρος, όπως σας είπα, της ομάδας υψηλού επίπεδου για την ισότητα των φύλων. Είναι Έλληνας, ανήκει στην πολιτική ομάδα της αριστεράς, την ΚΟΕ. Κύριε Παπαδημούλη, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα ξανά. Η δουλειά που κάνετε συνδέεται με αυτά που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ισότητα των φύλων και την ισόρροπη εκπροσώπηση. Έχετε το λόγο. Θα μιλήσει ελληνικά ο κύριος Παπαδημούλης, άρα βάλτε τα ακουστικά σας. First of thank you very much for your presence. Um... Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ε, εδώ θα χρησιμοποιήσω το δικαίωμά μου να μιλήσω στη μετρική μου γλώσσα ώστε να μπορέσω πιο ελεύθερα να εκφράσω όχι μόνο μια γραφειοκρατική προσέγγιση, αλλά και τα αισθήματά μου. Με χαρά να σας καλωσορίσω εδώ. Ε, βλέπω ότι μεγάλη πλειοψηφία όσων συμμετέχουν στο σεμινάριο είναι γυναίκες ε, και γι' αυτό θέλω να ξεκινήσω με μια εισαγωγική παρατήρηση. Η υπεράσπιση της ισότητας των φύλων είναι υπόθεση κατά τη γνώμη μου και των ανδρών και των γυναικών γιατί είναι διεκδίκηση βασικού ανθρώπινου δικαιώματος. Φυσικά στην πρωτοπορία αυτών των διακδικήσεων βρίσκονται γυναίκες φεμινίστριες, αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο ο στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε και να πείσουμε όλο ένα και περισσότερους άνδρες, έτσι ώστε να φτιάξουμε τις ευρύτερες δυνατές πλειοψηφίες ή δυνατόν και ομοφωνίες που να πιέζουν τα πράγματα προς τα μπρος. Ε, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μου ανέθεσε την τιμή και την ευθύνη να προεδρεύω σε αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου για τα θέματα της ισότητας και της διαφορετικότητας. Η ομάδα αυτή αποτελείται στη μεγάλη της πλειοψηφία από γυναίκες και από την αρχή της δράσης μας θελήσαμε να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο δράσης για την πενταετία που σε λίγο ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση θητείας του Ευρωκοινοβουλίου. Ένα roadmap με στόχους. Να δούμε πού βρισκόμαστε, πόσο απέχουμε από τους στόχους της πλήρους ισότητας και να επιδιώξουμε να κάνουμε βήματα για να μειώσουμε αυτή την απόσταση που χωρίζει την πραγματικότητα από τους στόχους μία μελέτη του ΟΗΕ, αν δεν κάνω λάθος, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αν συνεχίσουμε να προοδεύουμε με τους αργούς ρυθμούς που σήμερα σημειώνονται για την επίτευξη του στόχου της ισότητας θα χρειαστούμε πάνω από 150 χρόνια, ίσως 186 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Στο διάστημα αυτής της τετραετίας στον τομέα ευθύνης του High Level Working Group που έχω την τιμή να προεδρεύω πετύχαμε κάποια πράγματα. Εγκρίναμε αυτό τον χάρτη πορείας, ομόφωνα. Τον εισηγηθήκαμε στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα και σε συνεργασία με την Επιτροπή Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαστε δύο ομάδες πίεσης που κάνουν ένα διαρκές lobbying για να κινηθούμε ταχύτερα. Αν δούμε την κατάσταση στο επίπεδο της πολιτικής εκπροσώπησης, θα δούμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την παρουσία γυναικών στην Προεδρία Πολιτικών Ομάδων ως πρόεδροι ή συμπρόεδροι σε αρκετές πολιτικές ομάδες σε επίπεδο ψηλότερο από ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών, με εξαίρεση την σκανδιναβικές χώρες όπου τα πράγματα είναι πιο μπροστά. Το ίδιο συμβαίνει και σε ό,τι αφορά στην Προεδρία Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που και εκεί έχουμε σημαντική γυναικεία παρουσία. Όταν ερχόμαστε τώρα στη διοίκηση του Κοινοβουλίου, Εκεί έχουμε κάνει μια σημαντική πρόοδο στο επίπεδο όμως του middle management, των head of units, της μεσαίας διοίκησης, όπου μέσα σε αυτή τη διάρκεια της θητείας, από τότε που θέσαμε τους στόχους, ανεβήκαμε από το 29% γυναίκες head of units στο 38% στις αρχές του 2019 είναι μια πρόοδος. Δεν είναι ικανοποιητική, αλλά είναι μια πρόοδος. Αν πάμε όμως να εξετάσουμε πώς είναι η κατάσταση στο επίπεδο των γενικών διευθυντών, στην κορυφή της ιεραρχίας, εκεί το ποσοστό της συμμετοχής των γυναικών είναι αρκετά κάτω από το 20% και δεν έχουμε κάνει πρόοδο. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε στην ιεραρχία της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο τα πράγματα για την εκπλήρωση της ισότητας των φύλων γίνονται και πιο δυσκολότερα και πιο αργά. Και άρα σε αυτό ε, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες, να αντιμετωπίσουμε στερεότυπα, ε, να επιταχύνουμε πορεία. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνουμε μια αξιολόγηση, ένα evaluation. Τι στόχους βάλαμε, τι πετύχαμε, πού θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, διότι θέλουμε να κληροδοτήσουμε στην επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, τα συμπεράσματα από το πώς υλοποίησαμε αυτό το χάρτη πορείας, φιλοδοξώντας η επόμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια για πρόοδο. Και θέλω να πιστεύω ότι στο Προεδρείο είτε στο τέλος του Μαρτίου είτε στις αρχές του Απριλίου που λύγει ε, η θητεία του Ευρωκοινοβουλίου θα ολοκληρώσει αυτή την αξιολόγηση με την ίδια ευρεία συνένεση που μέχρι τώρα ε, έχουμε πετύχει ε, να λειτουργούμε σε αυτά τα θέματα. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα στα οποία πήραμε πρωτοβουλίες και κάναμε βήματα. Ορισμένα από αυτά ο κ. Ντούκ τα ανέφερε ε, επιγραμματικά. Αναθεωρήσαμε την, ε, τις εγκυκλίους και τις οδηγίες που δίνονται προς όλες τις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου όσον αφορά στην ουδέτερη ως προς το φύλλο γλώσσα ή ως την ευαισθησία σε ό,τι αφορά την ισότητα στη χρήση της γλώσσας σε σχέση με το φύλλο. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, υπηρεσίες που συνεργαστήκαμε γι' αυτό, δεν είναι μία οδηγία μόνο προς τους διερμηνείς, είναι υποδείξεις, ιδέες, πρακτικά εφαρμόσιμες με παραδείγματα για τη λειτουργία όλης της διοίκησης και θέλουμε σε αυτό το θέμα ως Ευρωκοινοβούλιο, επειδή είμαστε ένα-δυο βήματα πιο μπροστά από άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς, να πετύχουμε και μια διοργανική συμφωνία. Δηλαδή αυτό που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Κομισιόν έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο και είμαι αισιόδοξο ότι θα προχωρήσει. Εμεί είμαστε ω Ευρωκοινοβούλιο πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά βρίσκουμε, να το πω, ανοιχτά αυτιά από την πλευρά της Κομισιόν. Δεν θα έλεγα το ίδιο πράγμα και για το Συμβούλιο. Χρειάστηκε στο Συμβούλιο πολλές φορές να στείλουμε και επιστολές διαμαρτυρίας γιατί χρησιμοποιούσαν μία πολύ μονόπλευρη ως προς το φύλλο υπηρεσιακή επίσημη γλώσσα. Μάλιστα εγώ κάποια στιγμή αναγκάστηκα να στείλω και γραπτή επιστολή στην ε, Προεδρία του Συμβουλίου και εισπράξαμε μια υπόσχεση ότι κάτι θα γίνει για να υπάρξει αυτή η διοργανική συμφωνία. Πιστεύω στη διάρκεια της επόμενης θητείας το νέο Ευρωκοινοβούλιο να κάνει βήματα σε αυτό. Ε, γιατί η η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά οφείλει να είναι πιο μπροστά. Θα ήθελα να κλείσω και με μερικά θέματα τα οποία είναι και λίγο πιο εχμηρά και που δεν αφορούν την τρέχουσα διοικητική λειτουργία. Σεξουαλική παρενόχληση. το συζητήσαμε με αφορμή αυτό το κίνημα του Me το οποίο απλώθηκε σε όλο τον πλανήτη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υιοθετήθηκαν ψηφίσματα με μεγάλη ε, πλειοψηφία και η ομάδα υψηλού επίπεδου της οποίας προεδρεύω οργάνωσε και μία ανοιχτή ακρόαση με τη συμμετοχή και εκπροσώπων του κινήματος Μητού και των αρμοδίων υπηρεσιών και των αρμοδίων διευθύνσεων για να ασχοληθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο ενεργά με αυτά τα θέματα. Να μην τα καλύπτει ένα πέπλο σιωπή και business as usual. Έχουμε κάνει κάποια βήματα. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κι άλλα. Και η ομάδα εργασίας της οποίας προεδρεύω ε, πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει μια δέσμευση και το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ξανασυζητήσει αυτά τα θέματα, έτσι ώστε τα βήματα που έχουν γίνει να συνεχιστούν και να βελτιωθούν. Ένα δεύτερο θέμα είναι η διακρίση σε βάρο των γυναικών στην αμοιβή της εργασίας. Δυστυχώς αυτό το pay gap δεν υπάρχει μόνο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντί να μειώνεται υπάρχουν κράτη-μέλη που αυξάνεται. Όπως επίσης δυστυχώς υπάρχουν και τα θέματα της βίας κατά των γυναικών και η κύρωση και κυρίως η εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Και λυπάμαι να πω ότι υπάρχουν ακόμη και τώρα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και κυρίως δεν την εφαρμόζουν, διότι ένα θέμα είναι η νομική κύρωση και ένα δεύτερο θέμα πιο σημαντικό είναι η εφαρμογή. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι σε δύο μέρες η αρμόδια μονάδα για την ισότητα των φύλων υπό την διεύθυνση του κυρίου Κνούτσεν και με την ευθύνη του κυρίου Ροσέτη οργανώνει μια ειδική εκδήλωση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αξιολογήσουμε τα βήματα που έχουν γίνει και το τι ακόμη πρέπει να κάνουμε και θα σας ε, συνιστούσα ε, και να συμμετάσχετε όσες και όσοι είστε παρόντες μεθαύριο εδώ στο Κοινοβούλιο και να πάρετε και ένα φυλάδιο το οποίο φωτογραφίζει, αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση με αριθμούς, με ποσοστά και με στοιχεία και με συγκρίσεις με το παρελθόν για να βλέπουμε και την πρόοδο που έχουμε κάνει αλλά και την απόσταση που μας χωρίζει από το στόχο της επίτευξης της πλήρους ισότητας που είναι προφανώς θέμα δημοκρατίας και αφορά εξίσου και τους άνδρες και τις γυναίκες. Σας ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας μείνουν ε, τα εξή ότι και οι άνδρες πρέπει να συμμετέχουν και εσείς είστε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Όταν έφτασα στις Βρυξέλλες ε, πριν από 15 χρόνια ε, ένας είπε ότι βαρέθηκα ε, γιατί οι γυναίκες ε, δεν καθαρίζουν πολύ καλά με τη σκούπα πίσω από το ψυγείο και θέλω να ασχοληθώ με αυτό τέλο πάντων πιο πολύ για πλάκα δηλαδή ασχολούνταν μετά των γυναικών. Τώρα πρέπει να ασχοληθούμε όμως σοβαρά με αυτά τα θέματα και με την ισότητα των γυναικών. Επίση, είπε ότι μέχρι τη μεσαία διοίκηση οι γυναίκε υπάρχουν και μετά η άλλη οροφή αρχίζει από τα πιο ψηλά κλιμάκια και πάνω. Σήμερα. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι άντρα, έτσι, ο Αντώνιο Ταγιάννη. Ο Ντόναλτ Τάσκ επίση είναι άντρα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόεδρο τη Κριτική Τράπεζα είναι άντρα. Ε, ο Ντέισε Μπλούμα είναι ο πρόεδρο. Α, δεν είναι. Δεν είναι άντρα! <laughs> λέει ο πρόεδρο του Eurogroup. Α, αντικαταστάθηκε. Αντικαταστάθηκε. Αλλά και αυτό άντρα είναι, μάλιστα, ναι. Και ο αντιπρόεδρο και Τράπεζα τράπεζας είναι άντρα. Ε, ανησύχησα όταν ε, κατάλαβα, νόμιζα ότι κατάλαβα ότι μου ότι ο Ντάσικλου δεν είναι άντρα και δεν το φανταζόμουν. Ανησύχησα μάλιστα, τέλο πάντων. Ο Καρ Χάιντ Λάμπερτ είναι στο, ε, δικαστή, στο ελεγκτικό συνέδριο. Λούκα Χαγιέρ, ή κάπω έτσι, και τέλο πάντων και άλλοι. Όλοι άντρε. Αν όμω κατεβαίνουμε, φτάνουμε στη μεσαία διοίκηση και δούμε ε, στις εκτελεστικούς οργανισμούς, για παράδειγμα, ποιοι είναι επικεφαλής, σε έναν οργανισμό ε, θα βρούμε μια γυναίκα. Έχουμε για την ασφάλεια των τροφίμων, την Ευρωπαϊκή Αρχή, έχουμε για τις μεταφορές, για τα χημικά, έναν οργανισμό. Έχουμε και έναν οργανισμό για την ισότητα των φύλων. Σε αυτό το επίπεδο θα βρει κάποιο γυναίκε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι ε, πίεσε τα άλλα θεσμικά όργανα για να προωθήσουν την ισότητα των φύλων. Είχαμε μάλιστα ακούσει πριν δύο-τρία χρόνια ε, και για το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι δεν έχετε μια γυναίκα που είναι εκεί που ε, ε, ρυθμίζονται οι νομισματικές πολιτικές και από τους 29 γενικούς συμβούλους επίσης δεν ήταν ε, σε δύο δεν ήταν ε, γυναίκα πουθενά και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απέτησε το Κοινοβούλιο χωρίς να συμβεί ε, όμως αυτό. Ε, το είπε Άγγελα Μέρκελ. Θα το λάβουμε υπόψη την επόμενη φορά. Uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν πριν φύγετε θα είχατε την καλοσύνη να απαντήσετε σε μια ερώτηση παραπάνω από μία. Πέντε λεπτά όμως έχουμε γιατί έχουμε αργήσει λίγο. Έχετε λοιπόν κάποια ερώτηση προς τον κύριο Παπαδημούλη και τον ε, Ζάουμε. Απλά πριν πάρετε το λόγο να μας πείτε δωματεπώνυμο και μέσο που εκπροσωπείτε. Και για το πλαίσιο της εξαρτίας μη ε, του, ίσως, αν θέλετε. Δεν έχει να ρωτήσει κανείς. Λοιπόν, 35 άτομα έχουν υπογράψει αυτή την εκστρατεία μη του κατά της παρενόχλησης. Ε, εδώ. Είστε αποχωρητευμένος. Περισσότεροι από 35 αυτοί που έχουν περάσει αυτό το training yeah. Ναι. είμαι ένας από αυτούς. Το βρήκα πάρα πολύ θετικό και με ενοχλεί ο μικρός αριθμός και είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι από τη νέα θητεία αυτό το training πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Και έχω την τιμή να έχω υπογράψει μια επιστολή ε, εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας μαζί με προέδρους άλλων τριών πολιτικών ομάδων από τους πράσινους, mm. τους σοσιαλιστές, τους φιλελεύθερους και την αριστερά, δηλαδή τέσσερις πολιτικές ομάδες, οι οποίες συνιστούν και την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίες ζητούν πρώτον να γίνει υποχρεωτική αυτή η εκπαίδευση mm. από την επόμενη θητεία. Δεύτερον, οι θεσμοί που έχουμε δημιουργήσει για να αξιολογούμε τις καταγγελίες για το harassment μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υφίστανται και μια εξωτερική αξιολόγηση από ανεξάρτητους ειδικού, έτσι ώστε να έχουμε τη βοήθεια των ψυχολόγων, των κοινωνιολόγων, αυτό που λέμε στην ευρωπαϊκή γλώσσα best practices και θέλω να πω ότι στο hearing που οργανώσαμε ως High Level Working Group είδα ότι για παράδειγμα το Βρετανικό Κοινοβούλιο έχει πολύ πιο προηγμένους θεσμούς και μια πιο προχωρημένη εμπειρία στο πώς αντιμετωπίζει καταγγελίες για, για harassment. Άρα, σε αυτό το τομέα νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα μπρος δυστυχώς αντιμετωπίζουμε αντιδράσεις από συντηρητικά στερεότυπα και από δεσποτικές αντιλήψεις παλαιών εποχών. Έχουμε και ευρωβουλευτές οι οποίοι βγαίνουν στην Ολομέλεια και λένε βεβαίως οι γυναίκες πρέπει να αμείβονται λιγότερο διότι είναι πιο κοντές, πιο αδύναμες, έχουν μικρότερη μυϊκή μάζα, μπορούν να προσφέρουν λιγότερο αυτό προκάλεσε αντιδράσεις όπως καταλαβαίνετε. Υπέστη και κάποιες κυρώσεις ο Ευρωβουλευτής που εκτόξευσε τέτοιες εκφράσεις οι οποίες παραβιάζουν και άρθρα του κανονισμού αλλά προσέξτε κάτι προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρώντας ότι του περιορίστηκε με το μικρό πρόστιμο που του επιβλήθηκε η ελευθερία της έκφρασης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαίωση. Άρα πρέπει να βαθύνουμε πολύ παραπάνω τη σκέψη μας γύρω από κάποια πράγματα που στην Ευρώπη τα θεωρούσαμε αυτονόητα. Αναδεικνύεται και το πρόσωπο μιας σκοτεινής Ευρώπης και το ζούμε σε πολλές χώρες. I don't, know. Δεν ήταν αστείο είπε αυτός ο άνθρωπος ότι είναι πιο κοντές οι γυναίκες, άρα πρέπει να μείβονται λιγότερο. Σαν αστείο ακούγεται, σαν ανέκδοτο. Αλλά ήμουν παρούσα και το άκουσα με τα αυτιά μου. Είναι αληθινή ιστορία, παρότι μπορεί να μας εκπλήσει. Δηλαδή, ε, ας το πάμε και πιο μακριά, ότι τα παντελόνια μιας γυναίκας, επειδή είναι πιο κοντά, να κοστίζουν και λιγότερο. Τέλος πάντων, επειδή ε, καθυστερήσαμε λίγο, σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Τώρα, ένα από τα αφεντικά των υπηρεσιών αυτών θα έρθει εδώ, η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων, που εδρεύει στο Βίλνιους της Λιθουανίας, θα έρθει εδώ. Βιργίνια Λαντμπακ λέγεται. Έχει παλαιά ιστορία εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ήταν και υπουργό εξωτερικών στην, της Σουηδίας. Χαίρομαι που ήρθες εδώ και που θα μας μιλήσει για τη δουλειά σου. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ενθουσιασμένη που έχω την ευκαιρία πριν τις εκλογές να σας μιλήσω για την εξουσία και να ξεκινήσω θέτοντας το ερώτημα ποια είναι η δική σας εξουσία. Εσείς θα είσαστε ένα δίμερο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν πάτε πίσω στη χώρα σας, ποια είναι τα πιστικά επιχειρήματα που θα μπορούσατε να πείτε στις γυναίκες αλλά και στους άντρες για να επηρεάσετε το εκλογικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς, Φαντάζομαι ότι ήδη οι εκλογικοί κατάλογοι, οι λίστε αυτέ είναι έτοιμε από τα κόμματα. Και επομένω δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη θέση που έχουν μπει διάφοροι υποψήφοι. Αλλά εσεί μπορείτε να επηρεάσετε την ψήφο των ανθρώπων. Μπορείτε να δώσετε επιχειρήματα. Γιατί αυτού του λίγους ή του πολλού ανάλογα με την ιδιαιτερότητα τη χώρα, αυτοί οι λίγοι, περιπτώσει, εκπρόσωποι του γυναικείου φίλου πρέπει να είναι εκεί. Θα σα δώσω κάποια επιχειρήματα για να δούμε τι μπορούμε να πούμε. Και συνεχεία μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί κάθε χώρα είναι διαφορετική, κάθε κουλτούρα είναι διαφορετική και άρα θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να επηρεάσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές πραγματικότητες. Πιάσαμε μια χρονιά, το 1979, για να σας δείξουμε πόσες γυναίκες είχαμε στο πρώτο Ευρωκοινοβούλιο που εξελέγει απευθείας από εκλογές. 17 100 είχαμε. 40 χρόνια μετά, να η αλλαγή που έχουμε, να η αύξηση που έχουμε. Είναι μεγάλη αλλαγή. Δεν έχουμε τις λεπτομέρειες αναχώρα, αλλά η γενική εικόνα ήδη σας δείχνει ότι πρέπει να δράσουμε. Και εδώ έχουμε το δίκτυ για την ισότητα των φύλων. Μπορείτε να μην ξέρετε τι κάνει η υπηρεσία μου. Έχουμε μια ιστοσελίδα, έχουμε και ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάρα πολύ ε, για να παρατηρήσουμε την ισότητα των φύλων και την πρόοδο αυτής της ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λέει λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι τομείς, ο τομέας εξουσίας, όχι μόνο η πολιτική εξουσία, όπου οι εκπροσώπηση των γυναικών είναι όλο και περισσότεροι, αλλά είναι από τις χαμηλότερες σε σχέση με άλλους. Και αυτό δείχνει το χάσμα. Αν πούμε, ας πούμε, το 100 σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Καμία διαφορά στο μισθό, η απόλυτη ισότητα σε όλα, ίση εκπροσώπηση γυναικών στις ε, ψηλές και μεσές και κατώτατες θέσεις. Και ένα είναι απόλυτη ανισότητα. Εμείς είμαστε στο μέσο περίπου για να φτάσουμε το 100, που θα ήταν 50% γυναίκες, 50% άντρες παντού. Πρέπει ακόμα να κάνουμε προσπάθεια για να, να τα καταφέρουμε. Να φτάσουμε στο 50. Απλώς. Αυτό είναι ο δείκτης του 2017. Φέτος, θέλω να σας, ενθαρρύνω να σας ενθαρρύνω να σας κοιτάξετε το φετινό δείκτη. Τον Οκτώβριο κάθε φορά κάνουμε τη δουλειά για να δούμε ποιος είναι ο δείκτης εκείνη τη χρονιά. Με, μέχρι τις εκλογές ε, η Ιταλία, ας πούμε, αύξησε την ε, εκπροσώπηση των γυναικών κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, γιατί έβαλε ποσόστοση. Και διάφορες άλλες χώρες είχαν πρόοδο. Θα σας πω ποια είναι η θέση της χώρας σας. Λοιπόν, στο κοινοβούλιο βλέπετε ότι στα εθνικά κοινοβούλια, ας πούμε, έχουμε 30% εκπροσώπηση των γυναικών. Οι γυναίκες υπουργοί είναι 30,5% που είναι ο μέσος όρος. Αυτό δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Ισπανία είναι εντυπωσιακή ε, περίπτωση όπου ο αρχηγός της κυβέρνησης είπε ότι θα έχει πολλές γυναίκες, θα τους δοθεί η θέση που τους αρμόζει και έχει πάρα πολλές γυναίκες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ε, μπορεί να μην συμφωνούν πολλοί άλλοι με αυτό, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε εκεί, σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, αν προχωρήσουμε. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Για τις ποσοστώσεις. Εννέα κρατημέλη έχουν εισαγάγει ποσοστώσεις στο εκλογικό του σύστημα και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Και τι συμβαίνει, βλέπουμε το Βέλγιο, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία. Είναι τα κράτη αυτά και παρακολουθούμε και αναλύουμε τι γίνεται σε αυτές α, τις περιπτώσεις. Μόνο η Κροατία, μία από τις εννιά, δεν αύξησε τον αριθμό των γυναικών για να υπάρξει ισορροπία. Όλοι οι άλλοι αυξήσαν τον αριθμό των γυναικών. Είσαστε υπέρ των ποσοστώσεων εγώ είμαι υπέρ του να συζητήσουμε το θέμα, να μιλήσουμε για την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Η ποσόστοση είναι μια ενδιάμεση λύση, θα λέγαμε. Υπό την έννοια ότι αναγκάζει τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, τους κέρβερους τροποντινά, αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, να αρχίσουν να ψάχνουν για τους κατάλληλους υποψηφίους και να ρωτάνε, ενώ έχουμε τα κριτήρια, έχουμε τις προϋποθέσεις για τις γυναίκες για να πάρουν αυτές τις α, θέσεις, γιατί δεν βάζουμε τέτοιες προϋποθέσεις για τους άντρες. Οι ποσοστώσεις μας δίνουν το έναυσμα για να σκεφτούμε. Και για τα μέσα ενημέρωσης τους δίνουν το βήμα για να θέσουν ερωτήματα και να ψάξουν να βρουν την αλήθεια. Να ένα επιχείρημα λοιπόν, οι ποσοστώσεις. Πρέπει να σκεφτούμε όμως αυτό δρομολογεί μια αλλαγή. Όταν συζητάμε τις ποσοστώσεις πολύ συχνά, όταν αρχίσουμε το ψάχνουμε α πούμε, τι βρίσκουμε. Βρίσκουμε το εξή. Γιατί οι γυναίκες, ακόμα και αν τους πλησιάζουν από τα πολιτικά κόμματα, γιατί οι γυναίκες, ακόμα και αν τους πλησιάζουν και τους προτείνουν θέσεις, αισθάνονται ότι δεν είναι έτοιμε και λένε όχι. Γιατί υπάρχει η κουλτούρα αυτή του μάτσο, ε, η ανδροκρατική κουλτούρα, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, και τμήμα αυτή τη ανδροκρατική λογικής είναι και παρενόχληση. Δεν, χρειάζεται κανεί να είναι θύμα προσωπικά της παρενόχλησης για να το καταλάβει. Πόσε γυναίκε στα εθνικά κοινοβούλια δεν μιλάνε για τον τρόπο με τον οποίο φύγεται η αξιοπρέπειά τους. Για τον τρόπο με τον οποίο υποτιμώνται. Ε, για τον τρόπο με τον οποίο δεν τις σέβονται. Ε, δεν εκτιμούν τις ε, ικανότητές τους. Όταν σκέφτεστε λοιπόν τις ποσοστώσεις, αθέλητα σκέφτεται κανείς ότι πρέπει να πάρει κάποια μέτρα για να αλλάξει η νοοτροπία και εδώ στο Κοινοβούλιο και αλλού. Και αυτό φέρνει και σκέψη για το τι άλλο πρέπει να γίνει. Τώρα, βλέπετε τη χώρα σας, στο, που είσαστε ακριβώς. Ήδη πριν 10 χρόνια συνέβη το εξής παράδοξο. Οι γυναίκες, οι νέες γυναίκες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όλο και περισσότερο ήταν απόφοιτοι από πανεπιστήμια. Και μάλιστα είχαμε περισσότερες γυναίκες απόφοιτους από τα πανεπιστήμια από τους άνδρες. Άρα θεωρητικά μπορούμε να πούμε, ναι, έχουμε μορφωμένες γυναίκες που μπορούν να πάρουν πολιτικά σωστέ αποφάσεις και μπορούν να επηρεάσουν ε, μια θετική εξέλιξη στην κοινωνία. Βλέπετε το 68% που είναι ο ευρωπαϊκός ε, μέσος Το 68% από αυτές ε, σπουδάζουν ε, κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, υγεία, τέχνες. Ξέρετε ότι αυτό σε αντιδιαστολή με την μηχανική τεχνολογία κτλ. Ε, είναι λιγότερο η επιστήμες του μέλλοντος. Επομένως, από τη μία έχουμε το δυναμικό που θα μας εξασφάλιζε είτε εδώ στο Κοινοβούλιο, είτε στις χώρες να εξασφαλίσουμε τη γνώση, να δώσουμε τη γνώση το τι πρέπει να αλλάξει για να γίνουν οι αλλαγές, για να κλείσει αυτό το χάσμα και να υπάρξουν μεγαλύτερες ευκαιρίες για τις γυναίκες. Αλλά οι γυναίκες αυτές, ενώ υπάρχουν, δεν χρησιμοποιούμε τις γνώσεις τους. Από την άλλη, έχουμε και το εξή δεδομένο, ότι οι γυναίκες δεν ασχολούνται, απαξιούν, γιατί δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις. Γιατί ας πούμε τα σχολικά προγράμματα είναι αυτά που είναι. Γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα σχολικά προγράμματα τόσο ώστε να προσελκύσουμε περισσότερα κορίτσια σε πολυτεχνικές σχολές ας πούμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο χάνουν ας πούμε και οικονομικά ωφέλη. Πέρυσι το μελετήσαμε και προέκυψε ότι θα ήταν μεγάλη ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη για την κοινωνία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κάναμε και ανακράτω μέλο, μάλιστα, αυτό. Το να κλείσουμε αυτά τα χάσματα. Αν βρίσκαμε έναν τρόπο να το πετύχουμε, θα βελτιώναμε και την οικονομία. Αλλά δεν το κάνουμε. Αυτό γιατί γίνεται λοιπόν. Γιατί η γυναίκα δεν ε, ασχολείται με την πολιτική ή γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε τι γυναίκε δηλαδή. Έχουμε το δυναμικό, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε. Είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Κοιτάξαμε και το ευρωβαρόμετρο και κάποια στοιχεία που μας δίνει. Πρόσφατα εκδόθηκε. Η συμμετοχή στην πολιτική συζήτηση είναι προϋπόθεση για να ασχοληθεί κανείς με την πολιτική. 40% γυναικών και 35% ανδρών, λέει ο ομιλήτρια, λένε ότι δεν ενδιαφέρονται. Θέλαμε να δούμε αν υπάρχουν διαφορέ στα νούμερα για τους νέους άντρες και γυναίκες ε, σε αντιδιαστολή με τους ε, ηλικιωμένου, ή μεγαλύτερους, για να το πω πιο ευγενικά. Τέλος πάντων, αυτό που βλέπουμε είναι ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να πούμε ότι πρέπει να έχει την εμπειρία, να κάνεις κάποια μαθήματα, να βρει τον τρόπο και τα κίνητρα για να ασχοληθεί με την πολιτική και το 45% των γυναικών δεν συζητάνε καθόλου πολιτική με κανένα. Τι σημαίνει αυτό. Ε, είναι και δικό σας ρόλος για να δρομολογήσετε αυτές τις συζητήσεις, για να ενδιαφερθούν οι γυναίκες για την πολιτική. Το σχολείο είναι ο ένας παράγοντας. Αλλά ο άλλος παράγοντας είναι τα ΜΜΕ που μπορούν να ενθαρρύνουν τις γυναίκες αυτές να συζητήσουν πολιτική. Να μην το ξεχνάμε λοιπόν και αυτό. Εδώ τώρα, στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό προκύπτει το δικό μας ίντεξ βλέπουμε τη χειρότερη διάσταση που μας ταλανίζει. Βλέπουμε Εδώ βλέπουμε την κατάσταση στην οικογένεια. Έχουμε τα παιδιά, ε, ίσως υπάρχουν και ηλικιωμένοι εξαρτώμενα πρόσωπα. Θα πρέπει να βοηθήσει κανείς τα παιδιά, ε, πρέπει να κάνει όλη αυτή τη δουλειά στο σπίτι και υπάρχει και μια συζήτηση για το ποιος κάνει τι, έτσι. Για την κατανομή των ρόλων, ας πούμε. Και όταν αναλύσαμε αυτό, είδαμε ότι πριν 10 χρόνια, συγκρίνοντας την κατάσταση ε, ανδρών και γυναικών, όπου ξοδεύουν τουλάχιστον μία ώρα τη μέρα στο σπίτι για αυτή την απλήρωτη εργασία, βλέπουμε ότι η δουλειά που κάνουν οι γυναίκες έχει αυξηθεί, Ε, και μόνο ο ένας από τους τρεις άνδρες ξοδεύει τουλάχιστον μία ώρα στο σπίτι για την οικογένεια. Μόνο ο ένας στους τρεις. Άρα δεν αλλάζει και τόσο η κουλτούρα και τα στερεότυπα για την οικογένεια. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι οι γυναίκες δεν έχουν χρόνο να ενδιαφερθούν ίσως για την πολιτική, για να κάνουν κάτι άλλο, να αναπτυχθούν προσωπικά. Δείχνει επίσης ότι και η πολιτική για να αναπτυχθεί χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται αφιέρωση αλλά πρέπει όλοι να μοιραστούμε και τα άχαρα καθήκοντα. Τι μας κρατάει πίσω. Λοιπόν, θύματα παρενόχλησης. Ε, ψηφιακά και μη ψηφιακά. Κάναμε μια μελέτη λίγους μήνες πριν και είδαμε ότι τα νέα κορίτσια αποφεύγουν να μιλήσουν. Γιατί όταν μιλάνε, τους κολλάνε μία ταμπέλα. Και η ομότιμή τους, αλλά και τα μέλη της οικογένειάς τους. Ε, όταν μιλάνε δηλαδή online, στο διαδίκτυο δηλαδή για την πολιτική. Οπότε αποφεύγουν. Κάναμε συνεντεύξεις με νέους ανθρώπους Υπάρχει, υπήρχε ένα κορίτσι, μια Σουηδέζα, που έλεγε ότι ό,τι και να πω, κανένα με ακούει. Μπορεί να συμβαίνει το ίδιο σε πολλές χώρες. Εμείς ε, ασχοληθήκαμε με 10 χώρες μόνο που τις αναλύσαμε πιο ενδελεχώς. Ετοιμάσαμε και την έκθεσή μας, είναι στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να τη διαβάσετε. Αυτό που είναι απογοητευτικό είναι η γενική στάση. Όχι μόνο η έλλειψη σεβασμού ή ο σεβασμός, αλλά το γεγονό ότι το να είσαι κορίτσι σημαίνει ότι εκ προημίου σε σέβονται λιγότερο. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν μιλούσαμε μόνο με σκληρά επιχειρήματα για λεφτά και τα λοιπά, θα αυξάναμε σαν γυναίκες την, το σεβασμό ας πούμε, που έχουν οι άλλοι για μας. Επίσης είπαμε ότι αν κλείσουμε το μισθολογικό χάσμα ή μάλλον το χάσμα που υπάρχει στις επιστήμες ε, και πάνε σε πιο θετικές επιστήμες. Αυτό θα επηρεάσει και το μισθολογικό χάσμα, θα επηρεάσει πολλά πράγματα. Αν είχαμε περισσότερες γυναίκες και αν αποφάσιζαν να αλλάξουν σε εθνικό επίπεδο τα κράτη-μέλη ε, αυτό το διαχωρισμό που υπάρχει στην εκπαίδευση, ήδη από εκεί θα είχαμε επιχειρήματα για να πάρουν και πιο πολλές γυναίκες στην πολιτική. Ένας Καναδός Πρωθυπουργό το 2015, όταν το ρωτήσαν, είπαν, είπε μάλλον ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, και η ώρα, το ρώτησαν γιατί. Γιατί φτάσαμε στο 2015, είπε. Ε, εμείς τι έχουμε να πούμε, ότι φτάσαμε ήδη στο 2019. Ένας λόγος περισσότερο για να δράσουμε τώρα. Πέρασαν 40 χρόνια και μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια γίνανε ελάχιστες αλλαγές, μικρές αλλαγές. Οι γυναίκες έχουν δυναμικό, είναι μορφωμένες, τα ΜΜΕ θα πρέπει να τις προβάλλουν αυτές τις γυναίκες. Θα πρέπει να κάνουμε σοβαρές δράσεις για να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. It's a... Πραγματικά είναι λυπηρό γιατί είναι τόσο δύσκολο να αλλάξουν τα παραδείγματα και τα μοτίβα ότι κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα στο σπίτι οι γυναίκες 17 με 36% μόνο η διαφορά από θαρρυντικό μέσα 40 χρόνια τι έχει αλλάξει Είμαστε λίγο πίσω στο χρόνο, αλλά παρόλα αυτά θα δώσω το λόγο σε όποιους θέλουν. Εσείς με το λευκό φουλάρι καταρχάς. Ευχαριστώ από την Κροατία γράφω για ένα πολιτικό ε, μαγκαζίνο. Αναφέρατε την Κροατία. Είναι μια από τις χώρες που έχει σαγάγει ποσοστώσεις. Θα ήθελα να πω ότι ο λόγος ε, για τους οποίους δεν έχουν αυξηθεί ε, τα νούμερα είναι ότι οι άντρες είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Τι κάνουν, να βάζουν 40% γυναίκες, 40% ενό από τα δύο φύλλα που πρέπει να είναι στον κατάλογο, εγώ παραδείγματο χάρη για τι βουλευτικέ, περιφερειακέ, δημοτικέ εκλογέ κτλ τις βάζουν μεν στον ε, κατάλογο, αλλά σε, χαμηλό, ε, σε χαμηλή θέση, όχι εκλέξιμη. Και το μόνο κόμμα που το άλλαξε αυτό, για πρώτη φορά θα το δούμε τώρα, είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που έχει βάλει ένα σύστημα, αν μπορώ να το πω, φερμουάρ, δηλαδή ένας άνδρας σε μια γυναίκα. Ουσιαστικά ε, τους επιβλήθηκε να το κάνουν αυτό για τις τελευταίες εκλογές μαζί με τους συντηρητικούς ε, πλήρωσαν πρόστιμα γιατί δεν είχαν αρκετές γυναίκες στο κοινοβούλιο. Και στις τελευταίες εκλογές ήταν λιγότερες οι γυναίκες από ότι τα τελευταία 20 χρόνια που εκλέγονται άμεσα. Έτσι. Άρα πάμε προς τα πίσω. Αυτό είναι το σχόλιο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Κροατία και αν έχετε συνομιλήσει με πολιτικούς εκεί. Απάντηση. Ναι. Πρώτα απ' όλα Μ' αρέσει πολύ να βλέπω τα σου ειδικά μέσα. Πριν τι εκλογέ πριν από λίγου μήνε. Γιατί τα μέσα, τα μίντια ε, έχουν την, το ρόλο του. Και σε πολλές συνεντεύξεις ε, ή debate δεν αναφέρεται η ισότητα των φίλων κτλ. Παίζετε κι εσείς λοιπόν ένα ρόλο ε, οι δημοσιογράφοι για να συζητηθούν αυτά τα θέματα, να προβληθούν περισσότερο. Και συνήθως επισκεπτόμαστε τα κράτη-μέλη και για την Κροατία κάποιος πήγε ή θα πάει τέλος πάντων από εμάς σύντομα και αν ναι θα έρθουν και σε επαφή μαζί σας σίγουρα. Άλλη ερώτηση εκτός μικροφώνου. Ε, ε, Είμαι από την Κροατία και εγώ. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα της ποσοστώσης, θέλω να προσθέσω κάτι ότι ακυρώνεται και το ψηφοδέλτιο σε περίπτωση που δεν ε, είναι σεβαστή η ποσόστοση. Αυτό είναι ένα μέτρο που θεωρώ ότι αν εφαρμοστεί θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Και σε ό,τι αφορά τα μίντια, υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι στι ευρωεκλογέ το 50% των υποψηφίων ήταν γυναίκε, πήραν όμω ε, μόνο 20% κάλυψη από τα μέσα ενημέρωση. Έτσι, προ ενημέρωσή κάποια στοιχεία. Hello, I'm... Γεια σας, από τη Ρουμανία είμαι τη χώρα που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου αυτό το εξάμεινο και έχει και πολλές ε, πολιτικούς, ε, η Πρωθυπουργό και πολλές υπουργοί είναι γυναίκες στη Ρουμανία. Μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες πραγματικά μπορούν να εργαστούν στον πολιτικό στίβο. Γιατί στη δική μου τη χώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι ναι μεν είναι στην εξουσία, έχουν ε, υψηλά αξιώματα, όμως ουσιαστικά ακολουθούν τις αποφάσεις που λαμβάνουν άντρες, άλλοι στην πολιτική. Απάντηση. Συνήθως, κοιτάξτε, ναι δεν μας εκπλήσει. Αυτά τα ερωτήματα μου τα θέτουν σε πολλές επαφές που έχω θα σας δώσω την προσωπική μου άποψη. Αν δεν υπάρχει μια κρίσιμη μάζα, είναι πιο δύσκολο για τις γυναίκες διότι εκφοβίζονται κατά κάποιο τρόπο και καλό να υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξης. Αν όμως ε, είμαι η μόνη γυναίκα γύρω από άνδρες, ε, δεν νιώθω συνήθως ε, τόσο πολύ δυνατή, ισχυρή. Οπότε, ακόμη και αν έχουμε, όπως στη δική σας περίπτωση, στην κυβέρνηση μια γυναίκα πρωθυπουργό και στη Λιθουανία η πρόεδρος της χώρας είναι γυναίκα. Δεν αρκεί όμως αυτό. Πρέπει να υπάρχει αυτή η κρίσιμη μάζα. Γι' αυτό μιλάμε για ποσοστώσεις, ε, γιατί συνεισφέρουν σε αυτό οι ποσοστώσεις. Πρέπει να στηρίξουμε τις γυναίκες που έχουν ήδη ε, κάποιο υψηλό αξίωμα, γιατί έτσι μπορεί κανείς να φέρει και την ποθητή αλλαγή. η γυναίκα μπορεί να εστιάζει και σε κάποια άλλα θέματα, τις πάνω μπορούμε να έχουμε μια ευρύτερη προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να γίνει να είναι απομονωμένη. Τελευταία ε, σε ερωτήσεις, πολύ σύντομα παρακαλώ. Ζούλια Μπλάζη, από την Ιταλία, η χώρα μου. Ποτέ δεν είχε πολλές γυναίκες, τόσες πολλές γυναίκες στη Βουλή. Και τώρα ε, υπάρχει κίνδυνος να περάσει μια πολύ κατασταλτική νομοθεσία. Δεν αρκεί να έχεις γυναίκες ε, ε, στη πολιτική, αλλά να είναι και φεμινίστριες. Αν μπορεί να γίνει κάτι στο πολιτιστικό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί η φαλοκρατική κουλτούρα. Αυτό είναι καλό και αυτό δεν λύνεται μόνο με τις ποσοστώσεις. Ε, πρέπει η δράση να γίνει σε βαθύτερο επίπεδο, πολιτιστικό επίπεδο. Δεν ξέρω αν αυτό προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κάποια υποχρεωτική εκπαίδευση, κάτι τέτοιο για να αντιμετωπιστούν στις ρίζες τους αφαλοκρατικά αυτά ε, φαινόμενα. Απάντηση. Νομίζω ότι και ο Αντιπρόεδρος Παπαδημούλης μίλησε για ουδέτερης προς το φύλλο γλώσσα ε, και θα σας ενθάρρυνα ε, να το δείτε, έχουμε ένα πάρα πολύ ε, χρήσιμο διαδραστικό εργαλείο για την ουδέτερη ως προς το φύλλο γλώσσα στην επικοινωνία. που κανείς να χρησιμοποιήσει τα mail του κτλ. Και κάτι άλλο, έχουμε και άλλα εργαλεία, μια εργαλειοθήκη διαδραστική στο διαδίκτυο για την εσωτερική αξιολόγηση μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό έχει να κάνει και με τη φαλοκρατική κουλτούρα, για ε, τα κρούσματα παρενόχλησης, ε, φαινόμενα που μπορεί να μην είναι ορατά αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν α, δοκιμαστικές περίοδοι, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη δηλαδή αυτή η δοκιμαστική περίοδος για αυτή την εργαλειοθήκη, δεν έχουμε ακόμη τα αποτελέσματα από όλα τα κρατημέλη. Η φιλοδοξία μας όμως είναι σε όλα τα κράτη-μέλη να γίνει αυτή η αξιολόγηση, διότι δείχνει στο εσωτερικό επίπεδο ότι είναι αυτό που λείπει. Είναι θέμα νοοτροπία κουλτούρας, περιβάλλοντος. Είναι η γλώσσα που φταίει. Πώς όλα ε, μετρούν, όχι μόνο η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ θετικό αυτή η εργαλειοθήκη. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι της συζήτησης, αυτό το πάνελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που είπε η κυρία Λάμπακ ε, συμπεριλάμβανε πολλές στατιστικές. Τσεκάρετε τις στατιστικές για τη δική σας χώρα, μια και είσαστε δημοσιογράφοι. Αντώνιο. αν ζητήσει κάποιο δημοσιογράφο αυτέ τι στατιστικέ που παρουσιάστηκαν τώρα από την κυρία Λάγκμπακ να τι δώσει. Θα μπορούσατε να απευθυνθείτε στον Αντώνιο. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για καφέ, 10 λεπτών. Μπορείτε λιγάκι να ξεκουραστείτε πηγαίνοντα να πάτε τον καφέ σα και να τον πάρετε και να γυρίσετε όμω. Να μην χαθείτε στου διαδρόμου. Έτσι, ένα μικρό ξεμούδιασμα. Πάρτε τον καφέ σας και πίσω πάλι.